Θα πρέπει προφανώ να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων. Αυτό αληθεύει. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επομένω, η υποστήριξη τη μεταρρύθμισης αυτή θα επιτύχει μόνο αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά και αν εξασφαλίσουμε επίση τη δραστηριότητα έρευνα και διάσωση που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και να κάνω μια έκκληση στο τέλο τη θητεία αυτή. Σα παρακαλώ πολύ, εκινήστε εκ νέου την επιχείρηση Σοφία και δώστε τι μεγαλύτερε δυνατότητε έρευνα και διάσωση. Ο κύριος Ράντεφ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησα την εντολή μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την εποχή εκείνη η όλη ιδέα θέσπιση ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνορεφυλακής και Εκτοφυλακή ήταν ένα πολύ ασαφέ και θεωρητικό σχέδιο. Θεωρούσαμε ότι θα έβλεπε το φω τη ημέρα το νωρίτερα το 2030. Είμαστε όμω πάρα πολύ αφελεί τότε, γιατί μέσα σε ένα χρόνο είδαμε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες να καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασχίζοντας τα εξωτερικά μας ε, σύνορα και οι τότε συνοριοφύλακες δεν ήταν σε θέση να διχειριστούν ένα τόσο ακραίο φαινόμενο. Έπρεπε λοιπόν επιγόντως να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και συνειδητοποίησαμε ότι ο χώρος Σέγγεν είναι πάρα πολύ σημαντικός και ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων. Συνειδητοποίησαμε τότε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των εξωτερικών της σύνορων καταρχάς και τέσσερα χρόνια αργότερα να που συζητάμε για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοροφυλακής και Εκτοφυλακής. Λέμε ότι θα εμπεριέχει και ένα μόνιμο σώμα με δύναμη 10.000 ατόμων. Συζητάμε επίση για τι νέε αρμοδιότητε του οργανισμού αυτού. Μα νομίζω ότι ο οργανισμό αυτό από μόνο του αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύη μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών, αν θέλετε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα άνθρωποι είναι στο κατάλογο για το KGDI. Θα ήθελα πραγματικά να δώσω σε όλους το λόγο, όμως σας παρακαλώ πάρα πολύ ε, να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό που θα σας δώσουμε, διότι στις πέντε ψηφίζουμε και υπάρχει άλλο ένα θέμα στη μέση διάταξη πριν. Οπότε σας ζητώ πολύ ευγενικά να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό της παρεμβάσης σας. Η κυρία Σρόιντοβα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόταση σχετίζεται με το με πολύ μεγάλο λάθος που έγινε το 2015-2016 όταν τα εξωτερικά σύνορα της Σέγγεν δεν προστατεύθηκαν καταλήλως και υπήρξε διέλευση έως και 2 εκατομμυρίων ανθρώπων μεταναστών και προσφύγων. Κάποιοι από αυτούς ήταν όντως πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις φρικαλαιότητες του. Όμως πολλοί από αυτούς δεν ήταν επιλέξιμοι για άσυλο και θα πρέπει να επιστραφούν. Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξωτερικά τη σύνορα για λόγους ασφαλείας. Όταν έχουμε εκατομμύρια ε, μετανάστες οι οποίοι περνούν τα σύνορα, τότε η αίσθηση για τις χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, μετά από τρία χρόνια ε, καλής λειτουργίας, η νέα αυτή υπηρεσία, λέει κυρία Πίκουλα, ε, ο κύριος Πίκουλα θα εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντό τη Σέγγεν. Καλωσορίζω λοιπόν την θέσπιση αυτής ε, της ε, ε, δύναμης είναι μια αντίδραση στους κινδύνους που υπάρχουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να εξετάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για την ε, χορήγηση ασύλου. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το χώρο Σέγγεν, έχει να κάνει και με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Είναι καλό ότι θα έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Στίβενς, η κυρία Στίβενς. Κυρία, κυρία Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, Πάντα είμαστε υπέρ του Frontex. Πρώτη φορά το 2016 ο Frontex ανέλαβε το καθήκον να παρεμβαίνει περισσότερο στις επιστροφές ε, μετά από απόρριψη ασύλου. Και τώρα ξανά υποστηρίζουμε τον Frontex. Γιατί πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Frontex έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής. Μπορεί να είμαστε αποτελεσματικοί μόνο με ισχυρά εξωτερικά σύνορα και εδώ θα μας βοηθήσει ο Frontex. Περισσότερο, περισσότερη πόροι, προσωπικό, θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα έτσι τις προκλήσεις. Ο Frontex θα πρέπει να δραστηριοποιείται και σε μη ε, κράτη-μέλη, ε, χώρες που βρίσκονται μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Frontex θα βοηθάει στις επιστροφές από το Μαρόκο, προς μια άλλη χώρα μη μέλος, την Νιγηρία για παράδειγμα, τον Νίγηρα. Αυτό δεν μπορούσαμε, δεν το κάνουμε. Είχαμε χάσει αυτή τη δυνατότητα στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Να ε, πω ότι λυπάμαι ότι σε σημαντικό θέμα που ε, χιλιάδες ζωές εμπλέκονται και εκατομμύρια ε, ευρώ ε, δεν ε, γίνονται τακτές οι ερωτήσεις και δεν γίνεται καλή συζήτηση. Η λύση είναι το κράτος δικαίου. Αν, ο κόσμος, ε, ε, αν κάποιος επιδιώξει να μπει στην Ένωση παράνομα, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός κανόνας που θα λέει «Παρακαλώ, λυπάμαι, πρέπει να πάτε πίσω». Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει και νόμιμη οδός για την ε, αίτηση ασύλου, γιατί όλα τα πολιτισμένα κράτη δέχονται το δικαίωμα του ασύλου για αυτούς που διώκονται. Το κράτος δικαίου είναι το βασικό. Τα 11 δις ευρώ και οι έξτρα πόροι και η γραφειοκρατία θα βοηθήσουν ε, ε, να λύσουμε το πρόβλημά μας, ε, ενώ ένας πρακτικός κανόνας θα ήταν καλύτερος. Μπόκοβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια συμφωνία όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, προκειμένου να έχουμε ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στην Ευρώπη και προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο χώρος Σέγγεν. Δυστυχώς όμως δεν αντιμετωπίσαμε έτσι τα πράγματα του 2015. Επιτέλους όμως, τρία χρόνια μετά, συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την παράτυπη μετανάστευση και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποια βήματα ακόμα. Η εντολή του Frontex θα πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, να μπορεί να περιλαμβάνει και τις επιστροφές από τρίτη χώρα προς τρίτη χώρα. Στη Σλοβενία το 2015 είχαμε σε καθημερινή βάση χιλιάδες διελεύσεις των συνόρων μας και είδαμε ότι η τάση είναι ανωδική και τους τελευταίους μήνες και δεν νομίζω ότι πρόκειται να τροποποιηθεί πολύ στο μέλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι έρχονται από τη Βοσνία ή τη Σερβία θα, μπορούν να, θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφονται χάρη στο Frontex. Ο κυριο Λόπεθ Αγγελάρ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι Ευρω... Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Ισπανός. Είναι πολύ καλή η στόχη ενό στόχου ελεύθερη ε, ελευθερία ε, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ε, ε, έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και σε αυτό θα μας βοηθήσει η ακτοφυλακή, η συνοριοφυλακή ευρωπαϊκή με μια ε, νέα δυνατότητα 15.000 ε, ε, ανθρώπους με σημαντική χρηματοδότηση. Εμείς οι σοσιαλιστές συνεισφέραμε στη βελτίωση του κειμένου με τροπολογίες για να μην υπάρξουν επιστροφές σε τρίτες χώρες και να το συνδέσουμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το χάρτη των Θεμελιών Δικαιωμάτων που ισχύει. Όμως, πρέπει να ξέρετε ότι είναι αρκετά πικρό, πικρή η τελική γεύση, διότι υπάρχει τελικά μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και λιγότερη στον ανθρωπισμό. Στα νότια σύνορα της Ένωσης βρίσκεται η Ισπανία ε, και το πακέτο για το άσυλο ε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Το κανονισμό του Δουβλίνου επίση είναι μπλοκαρισμένο στο Συμβούλιο. Αυτά μένουν να γίνουν από το επόμενο Κοινοβούλιο. Ο κ. Μαριά έχει το λόγο, παρακαλώ. για άλλη μια φορά θέλω να μεταφέρω την κραυγή αγωνίας των κατοίκων των νησιών του αιγαίου για τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές και κυρίως το μεγάλο αριθμό παρανόμων μεταναστών οι οποίοι εισραίουν στην ελλάδα. πρόσφατα έγινε και εκδήλωση διαμαρτυρίας στην σάμο γιατί πλέον οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. πιστεύω ότι ο ρόλος της frontex πρέπει να βελτιωθεί να μπορέσει πραγματικά να κάνει σοβαρή δουλειά στα θέματα που αφορούν τη φύλαξη των συνόρων όχι μόνο στα θαλάσσια σύνορα γιατί βλέπουμε πλέον μεγάλη έλευση και από την μεριά των χερσαίων συνόρων την περιοχή του εύρου. επομένως εδώ πρέπει να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη βελτίωση της δουλειάς που κάνει η ίδια η frontex αλλά και στην περιοχή της Υπήρου που υποτίθεται υπάρχει η frontex στα